<laughs> Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Έχουμε τις ψηφοφορίες. Πρώτα. Ο πρόεδρος Μπούσεκ πάντα λέει ότι πρέπει να κάνουμε ένα τεστ στην αρχή πριν ψηφίσουμε. Ελπίζω να έχετε φέρει τις κάρτες σας, οπότε να κάνουμε ένα τεστ, μια δοκιμή Το ερώτημα είναι είστε έτοιμοι για τα Χριστούγεννα. Α, κάποιο θέλει να με παρέμβει τη διαδικασία. Ναι, δεν έχω την κάρτα μου, αλλά κάποια στιγμή θα την λάβω. Εντάξει, θα σε συμπεριλάβουμε, Πολ. Λοιπόν, κάντε μια δοκιμή για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αν είστε έτοιμοι για τα Χριστούγεννα είναι το ερώτημα. Τη δοκιμή βέβαια. Αρκετοί είναι έτοιμοι, βλέπω, για τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε με την πρώτη ψηφοφορία σχέδιο γνωμοδότησης ε, προς μια ψηφιακή στρατηγική. Ο κ. Και ο κ. Μπουτικόφερ είναι ο εισηγητής. Πρώτη γνωμοδότηση υπέρ, πρώτη μάλλον τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές να το επαληθεύσουμε παρακαλώ. Τροπολογία υπαρθμών 9. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές Λοιπόν, να απολυθέσουμε το δεύτερο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Μπορείτε να μετακινηθείτε δίπλα μήπως λειτουργήσει εκεί. Πάντως είναι σαφής πλειοψηφία τους, ή άλλος ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να το επαληθεύσουμε. Τροπολογία 21 λοιπόν, η ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται σαφώς. 22 υπέρ, κατά αποχές να το επαληθεύσουμε και αυτό. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν για το 22. Άρχιτη ψηφοφορία. της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24, 34 συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10, ε, μάλλον 50, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, όχι, θα πρέπει να το παληθεύσουμε. Τροπολογία 50, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Τροπολογία 47, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Άρχιτη ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Ε, συγχαρητήρια στον κύριο Μπουτικόφερ. Σημείο 5 της μέσης διάταξης τώρα. Πρόταση του Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωσης και τη Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου για την ε, εταιρική σχέση πρίμα. Η συγγήτρια είναι η κυρία Σακοράφα. Θα γίνει ε, ονομαστικά η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Σημείο 6, πρίμα και πάλι, με την Αλγερία αυτή τη φορά. Η συγγήτρια και πάλι η κυρία Σακοράφα. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Πέρας οφορίες. Εγκρίνεται. Σημείο 7. Πρίμα με το Λίβανο. Κυρία Σακοράφα και πάλι. Ηλεκτρονική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. Σημείο 8. Πρίμα με, την, με το Βασίλειο της Ιορδανίας. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά με ονομαστική κλίση. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τέλος έχουμε το σημείο 9. Διορισμό εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργεια. Ηλεκτρονικά θα γίνει ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και δεύτερη, Μπρίτα Τόμψον, ως ε, ε Αναπληρωματικό μέλος, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Η έγκριση των υποψηφίων. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Χέρτσοκ είναι εδώ, εκτό γνωρίζω. Σας συγχαίρουμε και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας για να μάθουμε τι κάνετε. Τέλειωσαν οι ψηφοφορίες και περνάμε στο επόμενο σημείο, σημείο 10 της μέρης σας διάταξης, επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, προετοιμασία της θέση του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020. Σχέδιο γνωμοδότησης ο κύριος Μαρινέσκου από το ΕΛΚ. Ένα λεπτό θα κάνουμε και θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα, το σημείο 10. Ένα λεπτό διαλυματάκι. Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, λείπει ο εισηγητή. Ένα εισηγητή, οπότε θα αλλάξουμε λίγο την ημερησία διάταξη. Θα πάμε στο 12 λοιπόν. Ενημέρωση σχετικά με τι ανεξελίξει διαπραγματεύσει για το EECC. Και για ο πρώτος τριμερή διάλογος έγινε την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου και σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μέχρι τον Απρίλιο του χρόνου το αργότερο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή για τον κώδικα επικοινωνιών. Κύριε Καστίγιο, κύριε Καστίγιο έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Περιγράψτε πολύ καλά την κατάσταση κύριε Πρόεδρε. Ο πρώτος τριμερής διάλογος έγινε στις 25 Οκτωβρίου, ο δεύτερος υπό την Εστονική Προεδρία πάλι. Θα λάβει χώρα το Δεκέμβριο, στις 6 Δεκεμβρίου. Πρέπει να πω ότι ο πρώτος τριμερής διάλογος διεξήχθη με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά ανταποκριθήκαμε σε μια ευρεία ε, πλειοψηφία που υποστήριξε μια εντολή στην Επιτροπή αυτή. Και τώρα για όσους γνωρίζουν καλύτερα, ε, κύριος σκοπός είναι να ενισχυθούν ε, οι επενδύσεις για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλή δυναμικότητας και για την ανάπτυξη του απαραίτητου περιβάλλοντος Τρία είναι τα κομμάτια φάσμα, πρόσβαση και υπηρεσίες. Κατά βάση. Ο επόμενος τριμερής διάλογος θα είστε στη... σε μεγάλο βαθμό στο κομμάτι του φάσματος. Θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα υπό την Εστονική Προεδρία. Θα ακολουθήσει η Βουλγαρία, η οποία συμμετέχει ήδη στους τριμερείς διαλόγους συντονισμός και η συμμετοχή όλων των ε, πολιτικών ομάδων μέσω των διαφορών σκιωδών είναι εξαιρετική. Δεν έχω να προσέψω τίποτα σε κανέναν. Σκοπός είναι να έχουμε τελειώσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Μόλις έχουμε ξεκινήσει, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για συμφωνία ακόμα, αλλά τα πράγματα βαίνουν καλώ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που το ακούω, ε, κυρία Καστήλιο. Και αναμένουμε να ακούσουμε τα όσα θα έχετε να μας πείτε μετά τους επόμενους τριμερείς διαλόγους. Σας ευχόμαστε καλή τύχη και καλή πρόοδο για αυτό το σημαντικό θέμα. Ευχαριστούμε. Πολύ ωραία. Προχωράμε λοιπόν τώρα στο σημείο 11 πηγαίνουμε αντίστροφα. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τι ευρωπαϊκέ στατιστικέ για τι επιχειρήσει. Ο εισηγητή μα είναι ο κ. Λεβαντόφσκι από το ΕΛΚΑ. Να πω πρώτα απ' όλα ότι λόγω του προβλήματος πληροφορική δεν έχουμε στη διάθεσή μας όλες τις γλωσσικές εκδόσεις του εγγραφού αυτού. Αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων σε αυτή την ε, ε, συνήθι νομοθετική διαδικασία. 15 λεπτά αφιερώνουμε σε αυτή τη συζήτηση να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε και τα 15 λεπτά, αλλά υπάρχει χρόνος εφόσον χρειάζεται. Κύριε Λεβαντός και έχετε το λόγο. Συγγνώμη, 50 λεπτά, όχι 15. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτό τον κανονισμό πλαίσιο για τα στατιστικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους ε, ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για στατιστικά δεδομένα υψηλής ποιότητας. Κάτι που διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται για τη μόνη πρωτοβουλία για θέματα στατιστικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στο Κοινοβούλιο έχουμε συζητήσει και για τη γεωργία και για τα κοινωνικά θέματα επίσης, για στατιστικά στοιχεία σε αυτούς τους τομείς. Καλωσορίζω αυτή την πρωτοβουλία. Ε, εντάσσεται στο REFIT, ε, καταργεί 10 σημαντικές πράξεις, τις οποίες αντικαθιστά με έναν κανονισμό και αυτό είναι πάρα πολύ καλό είναι ευπρόσδεκτο διότι σημαίνει ότι απλοποιούμε, απλουστεύουμε τα στατιστικά για τις επιχειρήσεις. Είναι όμως και μια πρόταση απαιτητική, ειδικότερα για όσους ε, συλλέγουν δεδομένα. Η συμφωνία πλαίσιο αφορούσε την απλούστευση, ε, την πιο συνεκτική προσέγγιση ε, όσον αφορά τα στατιστικά για τις επιχειρήσεις αλλά και την επέκταση στις υπηρεσίες σε τομείς ε, που δεν καλύπτονταν μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής τα στατιστικά για τις επιχειρήσεις αφορούσαν τη μεταποίηση κυρίως ενώ υπάρχει σαφής ανάγκη επέκτασης και στις υπηρεσίες. Εγώ συνομίλησα όχι μόνο με τους σκιώδεις συζητητές αλλά και με τους ενδιαφερομένους. Και φυσικά οι πιο ευχαριστημένοι είναι οι τελικοί χρήστε, διότι αυτοί έχουν μεγάλη ζήτηση στατιστικών στοιχείων υψηλή ποιότητα. Για του υπόλοιπου ενδιαφερομένου, αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτό που ονομάζουμε ε, ουδετερότητα του κόστου ή μάλλον εξοικονόμηση κόστου, ώστε να είναι το εγχείρημα αυτό πραγματικά αποτελεσματικό όσον αφορά το κόστος ε, να αντιστοιχεί στον ορισμό REFIT. Ε, συμφωνώ λοιπόν με την Κομισιόν ε, εδώ ουσιαστικά αναφέρομαι στην πρωτοβουλία για τη Eurostat. Ε, στην, ε, η πρωτοβουλία αυτή είναι της Eurostat ουσιαστικά. Εγώ προτείνω 27 πρωτο, τροπολογίες οι οποίες καλύπτουν τομεί. όπως κάποια περιορισμένη προσθήκη θεμάτων για στατιστικά στοιχεία, της κατεξοδότηση εκτελεστικές πράξεις, την έναρξη της περίοδου αναφοράς και το τέλος της. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες σήμερα, διότι είναι τεχνικές αυτές οι λεπτομέρειες, πιθανές επιπλέον δαπάνες και διοικητικός φόρτος και αυτό είναι σημαντικό για μένα ώστε να μην είναι υπερβολικός ο φόρτος, ειδικότερα για όσους ε, ε, συλλέγουν ε, τα δεδομένα. Η ασφάλεια των δεδομένων φυσικά είναι σημαντική και οι νέες μέθοδοι επίσης είναι σημαντικές με σκοπό το χαμηλότερο κόστος. Κάτι πολύ σημαντικό ειδικότερα όσον αφορά την εξοικονόμηση κόστους και τη φιλικότητα προς τους χρήστες. αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θέλω να επεκταθώ πολύ σε αυτή την πρώτη συζήτηση. Ας διαβουλευτούμε, ας διαπραγματευτούμε με τους κοιόδης συζητητές και αναμένω να ακούσω τις απόψεις τους, αλλά για μένα αυτό που είναι σημαντικό είναι να ανταποκριθούμε στη σαφή ζήτηση για στατιστικά στοιχεία υψηλής ποιότητας. Ε, στοιχεία που να είναι φιλικά προς το χρήστη και να αντιστοιχούν σε ένα εγχείρημα ρέφιτ πραγματικά. Ευχαριστούμε κύριε Λεβαντόφσκι. Στρέφουμε τώρα στους Κιώδης, εκ μέρους του Άλντε. Έχουμε τον κύριο Τελίτσκα. Παρακαλώ, Παύλ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Σταυρός Κυπέρ θα είναι σύντομο ε, και εγώ μπορώ να, να είμαι ακόμα πιο σύντομο και για πολύ καλό λόγο. Διότι η προσέγγιση μου ταυτίζεται απόλυτα με αυτή του εισηγητή. Μια πολύ λογική προσέγγιση που βασίζεται στα σωστά κριτήρια, στις σωστές αρχές. Συμφωνώ με τον κ. Λεβαντόφσκι επίση ω προς το ότι μπορούμε να ευθυγραμμιστούμε με τους στόχους ε, και με τις προτάσεις ε, της Κομισιόν επί της αρχής. Ταυτόχρονα υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Ένα από αυτά έχει να κάνει με την αξιολόγηση αντικτύπου. Θα πρέπει να είναι κάπως πιο πιστική η μελέτη αντικτύπου σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις. Και ιδιαίτερα σε αυτό που είπε ο κ. Λεβαντόφσκι οι επιπτώσεις ε, για τις επιχειρήσεις όχι μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ούτε η πρόταση όμως ούτε η μελέτη που είναι, είναι πιστικές σε ό,τι αφορά το κατά πόσο συμμορφώνεται αυτή η πρόταση με, την, ε, με το εγχείρημα Refit. Το πεδίο πάντως είναι σωστό οι τροπολογίες μου θα αφορούσαν ε, αυτά τα ζητήματα τα οποία ανέφερα. Βεβαίως είχαμε, ήρθαμε σε επαφή με τους διάφορους εμπλεκόμενους και οι περισσότερε τροπολογίε που θέλει να υποβάλει ο κ. Λεβαντόσκι είναι αυτές που θα επέβαλα και εγώ. Οπότε νομίζω ότι ε, υπάρχει σημαντική σύγκληση. Οι στόχοι είναι οι ίδιοι και κατά τη γνώμη μου μπορούμε έτσι να βελτιώσουμε αυτή την πρόταση. Κατά τα λοιπά, να μην επαναλάβω αυτά που είπε ήδη ο κ. Λεβαντόφσκι, για να μην χαθεί χρόνο να σα πω ότι σε ό,τι αφορά την πρώτη συζήτηση, η προσέγγιση του εισηγητή είναι τέτοια που ε, με κάνει να είμαι αισιόδοξο ε, για τη συνέχεια. Συμφωνώ με την προσέγγιση αυτή, συμφωνώ με την συντηρητική πλειοψηφία των ε, τροπολογιών, θα βρεθούν και συμβαστικέ τροπολογίε φαντάζομαι και είμαι βέβαιο ότι η πρόταση τελικά θα είναι καλύτερη. Δεν θα αναφερθώ στου τεχνικού ε, διακονισμού. Αυτά θα τα δουν οι εισηγητή με του και οι εισηγητέ. Ευχαριστώ τον κύριο Τελίτσκα. Ε, δεν ξέρω αν θέλει κάποιο άλλο το λόγο για αυτό το θέμα. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέλει να παρέμβει για αυτό το φάκελο. Ναι, Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Βεβαίω η Κομισιόν καλωσορίζει το πρώτο σχέδιο του εισηγητή του κ. και το πρώτο σχέδιο γνωμοδότηση. Ε, εκτιμούμε ιδιαίτερα την πραγματογνωμοσύνη του στο θέμα αυτό. Η έκθεση δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για αυτή την πρόταση και την επικοδομητική προσέγγιση που έχει ακολουθηθεί. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι η έκθεση είναι σε καλά χέρια αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες σε πολιτικό επίπεδο ε, ε, και ευχαριστούμε την Επιτροπή Ήτρε που μας δίνει την ευκαιρία να διευκρινίσουμε κάποια από τα ζητήματα αυτά. Ο στόχος της Κομισιόν με τον κανονισμό αυτόν, τον κανονισμό FRIPS, ε, είναι, οι στόχοι μάλλον είναι πολυσχηδείς, αλλά οι βασικοί ποιοι είναι. Πρώτον, να δώσουμε επιτέλους μια απάντηση στις ανάγκες των χρηστών δεδομένων όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να μειώσουμε το άθος των επιχειρήσεων. Δεύτερον. Τρίτον, μεσομακροπρόθεσμα ε, να έχουμε ένα στοιχείο ευελιξίας που να μας επιτρέπει να είμαστε επίκαιροι και στη συνέχεια. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά δυναμικά στατιστικά στοιχεία όπως ε, τα ICT, R&D, αλλά και την κοινοτομία. Χωρίς ευελιξία, χωρίς αυτή την ευελιξία, δεν θα μπορέσουμε να συνοδεύσουμε τις εξελίξεις στον οικονομικό τομέα. Μια σειρά από τροπολογίες που υπέφαλε ο εισηγητής, ε, εκ πρώτης όψεως, ε, μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι εύκολο να τις αποδεχτούμε, όμως θα πρέπει να διευκρινιστούν κάποιες από τις τροπολογίες αυτές, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε καταλάβει το ίδιο πράγμα. Ποιος είναι ο στόχος, είπα των τροπολογιών αυτών. Κάποιες από τις προτινόμενες τροπολογίες, ε, εφόσον τις έχουν καταλάβει καλά, οδηγούν στο ότι δεν θα μπορεί να πετύξει τους στόχους τη ε, αυτή η πρόταση. Θέλουμε λοιπόν εδώ να διευκρινίσουμε ε, τις προτάσεις της Κομισιόν σε ό,τι αφορά κάποιες τροπολογίες όπου εμείς έχουμε ανησυχίες. Η πρώτη τροπολογία και η πιο σημαντική για μας έχει να κάνει με την τροπολογία 28 στο παράτημα 2. Εκεί γίνεται αναφορά στην περιοδικότητα ε, των ε, τιμών των αποτελεσμάτων και της απόδοσης για τις, για τις μας στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων. Θέλω εδώ να διευκρινίσω ότι αυτές οι ανησυχίες ε, είναι, αφορούν μεταβλητές, ε, οκτώ μεταβλητές, οι οποίες απαιτούνται μηνιαίως. Από αυτές τις μεταβλητές μόνο δύο είναι καινούριε. Οι έξι προηγούμενες ήδη δίδονται τα στοιχεία αυτά μηνιαίως. Η τροποποίηση λοιπόν αυτή η τροπολογία οδηγεί στην πρώτερη κατάσταση. Από σε ό,τι αυτές τις δύο νέες μεταβλητές που είναι ο δείκτης ε, τζίρου, ε, κύκλου εργασιών για τις υπηρεσίες μεταξύ άλλων, πρέπει να πω ότι πάνω τα μισά κράτη-μέλη ήδη χορηγούν αυτά τα στοιχεία. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό αίτημα της Ευρωπαϊκής, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τράπεζας. Από το 2000 το ζητάει. Είναι σημαντικό για να μπορέσει να κάνει προβλέψεις για το ΑΕΠ, ε, για την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής νομισματικής Πολιτικής να έχει αυτά τα στοιχεία η ΕΚΤ. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ σε μια άλλη τροπολογία, τις τροπολογίες μάλλον 15 και 16. Αυτές οι τροπολογίες έχουν να κάνουν το μητρό του Eurogroup και την πρόταση της Κομισιόν κάποια άτομα στις Εθνικές Αστικές Αρχές που εργάζονται στην παραγωγή αυτού του μητρώου να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα για όλες τις πολυεθνικούς, πολυεθνικούς ομίλους ε, και για τις ξένες ε, νομικές αρχές. Αυτοί οι στατιστικολόγοι, αυτή η υπάλληλοι υπόκειται σε πολύ αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας και είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό, διότι ένας, ένας στατιστικολόγος, ένας, ε, ένας μέρος μιας στατιστικής υπηρεσίας θέλει να βάλει μια νομική μονάδα σε ένα ολόκληρο όμιλο να την τοποθετήσει εκεί που πρέπει, πρέπει να έχει μια σφαιρική εικόνα. Ιδάλλως ε, δεν θα ξέρει εάν αυτή η νομική μονάδα ανήκει στον τον όμιλο. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν έστω και ένα μικρό αριθμό ανθρώπων να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία αυτή. Πάντα βέβαια στα πλαίσια των κανόνων εμπιστευτικότητας που θα πρέπει να τηρήσουν. Τέλο, θα ήθελα να αφαιρθώ στην τροπολογία 22 που σχετίζεται με τη διεθνή, τα στατιστικά μάλλον ε, για το διεθνές εμπόριο ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τους τρόπους ε, διανομής. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν συλλέγονται. Υπάρχει όμως πολιτική πίεση για να προκύψουν τέτοια στοιχεία. Η ρητή αναφορά αυτών των στατιστικών στοιχείων ε, αναφέρεται στις, ε, στις πιλωτικές μελέτες και ε, θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα να, παράγει τέτοια στοιχεία, διότι είναι κάτι που ζητούν οι πολιτικοί θύνοντες. Το να διαγράψουν αυτή την αναφορά, όπως προτείνετε εσείς στην τροπολογία επαρθμών 22, δεν θα δώσει το κατάλληλο μήνυμα. Οι τροπολογίες 8, 9 και 10 τώρα ε, θέτουν κάποια θέματα τα οποία είναι τεχνικής υφής όμως και χρήζουν άλλου τύπου εξήγηση, πιο μακροσκελού και με γραφήματα. Ε, για αυτή την προκαταρκτική φάση της έκθεσης νομίζω πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, όμως ε, η Κομισιόν είναι απολύτως διατεθειμένη να διευκρινίσει σε μια τεχνική συνάντηση, αν θέλετε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, τα όποια ζητήματα ακόμα υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο ξανά στον κύριο Λεβαντόφσκι για τα ε, τελευταία του σχόλια. Παρακαλώ, Γιάννος. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που ακούω ότι συμφωνούμε και η προσπάθειά μου είναι να υπάρξει μια πραγματική ε, διαδικασία refit. Ε, έτσι λοιπόν σκοπός όλων μας είναι να μειώσουμε το άχθος για όλους ε, τους φορείς συλλογής στατιστικών ε, δεδομένων. Θεωρώ και εγώ ότι η στατιστική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμβαδίζει με τη ζωή των επιχειρήσεων, αλλά πρέπει να βρεθεί και μια ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία και την προβλεψιμότητα ε, για τις επιχειρήσεις. Για τα συγκεκριμένα θέματα που τέθηκαν σήμερα, ναι, πραγματικά επαναρχόμαστε σε τριμηνιές ε, περιόδους ε, συλλογής πληροφοριών για τις ε, τιμές. Ωστόσο, πρόκειται για μια διαδικασία ποσόστοσης. Σε κάποιες χώρες μηνιαίως ε, συλλέγονται αυτά τα δεδομένα. Σε κάποιες χώρες καταλαβαίνω όπως ε, στην Πολωνία αυτό δεν είναι πρόβλημα, σε άλλες χώρες όμως είναι πρόβλημα. Όσον αφορά την πρόσβαση, την πρόσβαση στα δεδομένα, η τροπολογία μου αφορά μόνο τις χώρες εκείνες όπου υπάρχει ήδη νομική ε, οντότητα για τα πιλωτικά προγράμματα με ενημέρωσε η Eurostat ότι έχουν ήδη συλλεγεί τα εμπορικά δεδομένα, οι στατιστικές πληροφορίες. Θα μπορούσα να συμφωνήσω κάτι τέτοιο να γίνει στο μέλλον, αλλά δεν ξέρω πώς σχετίζεται αυτό με τη σημερινή μας συζήτηση. Αυτό που κρατώ είναι ότι χαιρετίζουμε την απλοποίηση, την απλούστευση, την, τον εξορθολογισμό, την κατάργηση των δέκα νομικών πράξεων και την αντικατάστασή τους με μία, αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και πρωτοβουλίες ε, στη δικές σας, στην ε, γεωργία και στις, και, στα, και στις κοινωνικές στατιστικές και δυστυχώς η πρόοδος που σημειώνεται δεν είναι παρκός, ε, ε, δεν είναι παρκής. Αντιθέτως φαίνεται ε, αυτές οι διαδικασίες να επιβαρύνουν ε, δυσανάλογα πολύ τα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν ε, να θέσουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας τη φιλικότητα προς τον, τη φιλικότητα προς τον χρήστη και ως πρώην επίτροπος νομίζω ότι έχουμε κάθε δυνατότητα να βρούμε συμβιβασμό. Ευχαριστούμε. Προθεσμία καταβολής τροπολογιών είναι 30 Νοεμβρίου 2017. Ευχαριστούμε κύριε Λεβαντόφσκι για τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Και τώρα, επανερχόμαστε στο σημείο 10 της σας διάταξης. Επόμενο ΠΔΠ, προτεμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Ο κύριος Ήλα, ε, από ό,τι βλέπω, είναι έτοιμος να πάρει το λόγο εκ μέρους του συντάκτη της γνωμοδότησης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρου του κ. Μαρινέσκου, ο οποίο δεν κατάφερε να παρευρίσκεται. Επιτρέψτε μου να δούμε εν συντομία την πολύ περιεκτική έκθεση του κυρίου Μαρινέσκου. Ουσιαστικά καλύπτουμε όλα τα ζητήματα πολιτικής ε, της ΙΤΡΕ που σχετίζονται με τον προπολογισμό ε, αφορά τη στρατηγική της βιομηχανικής πολιτικής, την εμβάθυνση της ενεργειακής αγοράς, ε, αναφέρεται στην ενιαία αγορά, στα εργαλεία της, ε, απαιτεί καλύτερο συντονισμό των μέσων, ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τεχνολογίες ενημέρωσης και επικοινωνιών, ενέργεια, υποδομές αναφέρεται στον ορίζοντα 2020, στο διαστημικό προϋπολογισμό και στο νέο εμφανιζόμενο ε, ευρωπαϊκό πρόγραμμα ε, άμυνας. Πώς μπορούμε λοιπόν να συμβάλλουμε εμείς ε, στον νέο προϋπολογισμό και θα μπορούσαμε ίσως να βρούμε και λίγο χώρο να τροποποιήσουμε την έκθεση για να πούμε ότι αναφερόμαστε σε ένα συγκεκριμένο νούμερο το 3% να ε, δέδεται στην έρευνα και στα 120 δισεκατομμύρια για το πρόγραμμα 9 ότι έχουμε αποφασίσει από κοινού ότι δεν θέλουμε το FC2 να πάρει χρήματα από τα προγράμματα έρευνας και κοινοτομίας. Θέλουμε να αναφερθούμε στο EIT, γιατί και αυτό είναι κομμάτι του προπολογισμού που η ΙΤΡΕ ε, πρέπει να εκφέρει άποψη. Θα αναφερόμαστε επίσης στο χάσμα καινοτομίας, ε, στις συνέργειες που απαιτούνται στο ρόλο των δημιουργικών και πολιτιστικών ε, τομέων και κλάδων. Επίσης, όσον αφορά τους κανόνες, θα αναφερόμασταν ε, στα μέσω των καποκοπής ποσών, στην ενιαίο έλεγχο και στο ότι θεωρούμε ότι το πρόγραμμα 9 πρέπει να βασίζεται σε επιχορηγήσεις ε, και όχι οι επιχορηγήσει να αντικαθίστανται από δάνεια. Αυτά θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να μπουν στην έκθεση του εισηγητή και αυτή θα, είναι και... θα προσθέσουμε επίσης και τη θέση του ΕΛΚΑ σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στους σκιώδεις. Ε, κυρία Βέρνερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δυστυχώς ο κύριος Γκάια ε, βρίσκεται στην ομάδα διαπραγμάτευσης για τον προπολογισμό του επόμενου έτους, γι' αυτό και σας μεταφέρω τι θέσεις του. Καταρχά να σας ευχαριστήσω κύριε Μαρινέσκου για την γνωμοδότησή σας για το επόμενο ΠΔΠ. Αναφέρθηκαν πολλά σημαντικά ε, θέματα από τον κύριο Μαρινέσκου, τα οποία υποστηρίζει ε, και ο κύριος, Γκάια, όπως είναι η υποστήριξη της ενεργειακής ένωσης, του χώρου έρευνας και η ψηφιακή ενιαία αγορά. Όπως και ο εισηγητής, ο κύριος Γκάια θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι η απαραίτητη χρηματοδοτική πόρη για το ΣΕΦ και για τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά προγράμματα. Ωστόσο, Υπάρχουν και ορισμένα σημεία τα οποία θα ήθελα να τονιστούν ο κύριος Γκάια. Η Κομισιόν πρέπει να επικεντρωθεί στην ε, απασχόληση και την ανάπτυξη και να επιμείνει σε αυτό το θέμα, όπως και στο προηγούμενο πι Οι σοσιαλιστές επίσης υποστηρίζουν την ε, ε, υποστήριξη πολιτικών γύρω από ζητήματα που σχετίζονται και με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως είναι η ενεργετική αποδοτικότητα. Πρέπει να συνεχιστούν πολιτικές αντίστοιχες ε, ενίσχυσης ε, των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο κύριος Γκάιερ επίσης υποστηρίζει να υπάρξει επαρκή χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών οργανισμών προκειμένου να μπορούν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. Ο κύριος Γκάιερ επίσης θέλει να ξανατονίσει ότι τα προγράμματα που έχουν ε, αποδείξει την αξία τους και την αποτελεσματικότητά τους ε, αλλά και τα ε, προγράμματα έτσι και το Ταμείο Άμυνα δεν θα πρέπει να υποστούν καμία μείωση τη χρηματοδότησή του. Επίση, πρέπει να διατεθούν νέα χρήματα για νέε πρωτοβουλίε. Αντίστοιχε τροπολογίε θα καταθέσει ο κύριο Γκάιερ, ο οποίο και προσβλέπει στην καλή συνεργασία με τον εισηγητή και με του υπόλοιπου σκιώδου εισηγητέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Βάρνερ. Εκ μέρους των φιλελευθέρων κύριο Στυλίτσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι υπόθηκαν ήδη πολλά. Έχουμε κάποιες βασικές αρχές τις οποίες έχει συμπεριλάβει στο κείμενό του ο εισηγητής σε γενικές γραμμές. Μια γενική παρατήρηση θέλω να κάνω που πιστεύω ότι μπορεί να μας καθοδηγήσει και στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ, αλλά και στον τομέα της χάραξης πολιτικής. Ο εισηγητής τόνισε ε, το ζήτημα της καινοτομίας και ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει μείωση των ε, χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020. Σωστό αυτό. Ωστόσο υπάρχουν όμως και κάποιες πολιτικές αλλαγές σε ορισμένα κράτη-μέλη. Υπάρχουν εντάσεις και υπάρχουν και φιλοδοξίες να αναθεωρηθεί στο μέλλον η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και όχι απαραίτητα σε θετική κατεύθυνση. Ε, και μια τέτοια εξέλιξη βεβαίως θα μπορούσε να πλήξει ε, πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωση στον τομέα τη καινοτομία και τη έρευνα. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το έχουμε κατά νου σήμερα αλλά και στο μέλλον. Η ίδια παρατήρηση ωστόσο ε, αφορά και το οικοσύστημα που έχουμε στην Ευρώπη. Πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε, να σταθούμε στον ε, ανταγωνισμό με τους βασικούς μας ανταγωνιστές στο μέλλον. Πρόκειται για ζητήματα χρηματοδότησης και πιστεύω ότι θα πρέπει στο μέλλον να ε, επικεντρωθούμε περισσότερο στη συγχρηματοδότηση και την ίδιο χρηματοδότηση σε συγκεκριμένα ε, έργα και σε συγκεκριμένους κλάδες, κλάδους όπου χρειάζεται ακόμα χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όμως σημαντικό να μην ξεχνούμε ότι η Επιτροπή Ήτρε ε, είναι αρμόδια και για ένα άλλο ζήτημα που αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο συγκεκριμένα. Και το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι πάντοτε τμήμα του οικοσυστήματος. Βεβαίω, αυτά που είπε ο εισηγητή δεν μπορεί κανεί να τα σχολιάσει αρνητικά. Ωστόσο, τονίζω από δική μας, από μας πλευράς ότι διανύουμε μια δύσκολη περίοδο αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα, μεγάλες πιέσεις θα αντιμετωπίσει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Υπάρχουν διάφοροι συγκριτικοί δείκτες οι οποίοι θα ε, εφαρμοστούν στο επόμενο, το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό και εμείς χρειάζεται να έχουμε μια πολύ συγκροτημένη αντίληψη για το πώς θέλουμε να χαράξουμε την πολιτική μας. Αυτά ε, θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθούν και οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις. Παρ' όλα αυτά ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή δεν, έχω κάποιες, ε, δεν έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά το κείμενο του εισηγητή. Ευχαριστώ τον κύριο Τιλίτσκα. Για τώρα οι πράσινοι έχουν το λόγο. Ναι, μπορώ να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο κύριος, ε, ο, ο Παύλ προηγουμένως μάλλον, λέει ο κύριος Τούρμες. Ε, εδώ υπάρχει ένα πολιτικό θέμα. Οι Βρετανοί φεύγουν. Ε, πολλά από τα ζητήματα λοιπόν που συζητούμε στην Επιτροπή Ήτρε θέτουν το ζήτημα από πού θα προέλθουν τα χρήματα. Η έκθεση του κυρίου Μαρινέσκου δεν λέει τίποτα για τους δύο σπόρους. Εάν δεν έχουμε νέους ιδίους πόρους, θα βρεθούμε στριμωγμένοι. Θα πρέπει λοιπόν και στην Επιτροπή Ήτρε να μιλήσουμε για τους ιδίους πόρους. Είναι δύο τομείς όπου πραγματικά θα υπάρξει και μεγαλύτερη ε, αξιοπιστία ε, στο ευρύ κοινό. Η Ευρώπη είναι αυτή που κατάργησε την περιαγωγή. Η Ευρώπη είναι αυτή η οποία οδήγησε σε ένα πιο φτηνό ίντερνετ. Να ζητήσουμε λοιπόν ένα μικρό τέλος για την κάθε επικοινωνία που να μας επιτρέψει στο μέλλον τα χρήματα αυτά να βελτιώσουμε ε, το ευρυζωνικό σύστημα και να μειώσουμε το κόστος για τους πολίτες. Ε, το ίδιο ισχύει η ηλεκτρική ενέργεια. Ε, εάν δεν έχουμε μια ευρωπαϊκή αγορά φυσικά φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φτάσουμε σε χαμηλές τιμές. Όταν οργανώνεται μια εσωτερική αγορά χωρίς σύνορα, τότε υπάρχει και μεγιστοποίηση και καλύτερη χρήση των πόρων μας. Πρέπει να δείξουμε ότι η Ευρώπη μειώνει το κόστος για τους πολίτες. Αν θέλουμε λοιπόν ε, να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή και εκεί θα πρέπει να το πούμε. Το θέμα τώρα του κλίματος, του περιβάλλοντος. Σήμερα τη Δευτέρα στη Βόνη, αρκετά κοντά, οργανώνεται ε, μία διάσκεψη κοπ, της κοπ στην Βόνη, ε, Φίτσι, Ευθυγράμμιση λοιπόν χρειάζεται, όπως είπε και ο κ. Μαρινέσκου, τώρα για τη βιομηχανική πολιτική. Χάρη σε πολλέ πρωτοβουλίε ε, και του κυρίου Έλεν και του Κάρλος Μέιδα, τώρα είμαστε πολύ καλύτερα. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη, τη startup, το ρίσκο, ε, στις επενδύσεις. Όμως για τα μεγάλα βιομηχανικά σχέδια, εκεί χρειάζονται πολλά χρήματα. Και εκεί έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα. Πώς να ανταγωνιστούμε την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί ο Άλαν Μάσκ μπορεί να ανοίξει ε, μια μεγάλη ε, εταιρεία, μια μεγάλη κατάσταση. Ε, γιατί έχει πίσω την Αμερικανική κυβέρνηση με εγγυήσεις. Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Ο κ. Μαρτινέσκου λέει κάποια καλά πράγματα από αυτού ε, στην έκθεση και θα πρέπει ενδεχομένω να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο για τι ανάσχημε πηγέ ενέργεια τώρα. Εάν θέλουμε ε, να μπορέσουμε πέρα από τα σύνορα να, έχουμε μια καλύτερη διαχείριση, τότε θα πρέπει να έχουμε, δώσουμε και κάποια, να κάνουμε κάποιε παραχωρήσει. Εάν πέρα από τα σύνορα μπορούμε να εργαστούμε για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, εάν μπορούμε να δώσουμε εγγυήσει για αυτέ τι επενδύσει. Ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό θα μειώνει το κόστος για όλους ε, και είναι ακόμα ένα στοιχείο το οποίο θα ε, προσθέσω στις τροπολογίες που θα υποβάλλω. Ευχαριστώ τον κύριο Τούρμες. Από την ΚΟΥΕ τώρα η κυρία Σακοράφα έχει το λόγο παρακαλώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή την αρχική προσέγγιση που έχει κάνει όσον αφορά τις, το κρίσιμο ζήτημα της προετοιμασίας των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, και να τονίσω ότι κατά την άποψή μου το επόμενο πλαίσιο θα πρέπει να έχει έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα με κοινωνικό πρόσημο και αναδιανεμητικό ρόλο τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και στο εσωτερικό τους. Αυτή η κεντρική πολιτική επιλογή θα πρέπει να έχει το προβάδισμα απέναντι σε κάθε πολιτική ε, προτεραιότητα που μπορεί να μπει, είτε πρόκειται για το αντίπαλο δέος της ανταγωνιστικότητας, είτε για κάθε νεοφιλελεύθερη έμπνευση εγχείρημα τύπου Ενεργειακής Ένωσης, ενιαίας ψηφιακής αγοράς ή ακόμα και της Ένωσης των Κεφαλαίων Παράλληλα με όχημα της δημόσιας επενδύσεις και το δομικό χαρακτηριστικό την πλήρη απεξάρτηση από την οικονομική διακυβέρνηση και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το νέο πλαίσιο θα πρέπει να απαλλαγεί από κάθε τιμωρητική και αντιαναπτυξιακή προϋπόθεση μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, η συγκυρία των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαιτεί πλέον μόνο ένα επαρκές μέγεθος δαπανών, αλλά μια γενναία αύξηση με κυρίαρχο μοντέλο προετοιμασία και διοίκηση των πόρων, την αποκεντρωμένη διαχείριση και τι συμφωνίε εταιρική σχέση, η κατανομή των πόρων θα πρέπει να στηριχθεί και σε συμπληρωματικού δείκτε κοινωνική πρόοδου, πέρα από του παραδοσιακού που αφορά στο ΑΕΠ. Οι επιχορηγήσει θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βάση τη χρηματοδότηση. Ο διευρυμένο πλέον ρόλο των χρηματοδοτικών μέσων όπως του εξαιρετικά αναξιόπιστου Ταμείου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις ή του νέου Ταμείου Στρατιωτικοποίησης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την στήριξη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας, λειτουργεί τελικά σε βάρος αξιόλογων προγραμμάτων, όπως είναι ο Ορίζοντας 2020 και το κόσμε και φυσικά στην ανάγκη την αναθεώρηση των προτεραιοτήτων θα τοποθετηθώ θετικά. Με μια προϋπόθεση. Κάθε τέτοια κίνηση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, και σε συνδυασμό με τι αποφάσει για την ενίσχυση μια συλλογισμένη ευελιξία. Πιστεύω όμω ότι ένα μόνιμο σύστημα κινητοποίηση πρόσθετων πόρων θα ενισχύσει την ικανότητα ανταπόκριση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στις νέε προκλήσει, καθώ και σε καταστάσει εκτάκτου ανάγκη, όπω αυτή που προέκυψε από την προσφυγική κρίση. Τέλο, υπενθυμίζω την σημασία τη παραπέρα συνολική απλούστευση και την έμφαση στην ποιότητα των έργων και όχι στην ψηφοθυρική απορρόφηση. Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή μου, κύριε συνάδελφοι, σας καλώ σε εγρήγορση, γιατί οι παράμετρος του Brexit και η θολή εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι κρίσιμοι παράγοντες για την διαμόρφωση του νέου πλαισίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς, οι Ευρωβουλευτές, είμαστε εδώ και πρέπει να διαδραματίσουμε ένα πολυεπίπεδο, ενεργό και δυναμικό ρόλο σε όλη την διαδικασία της διαπραγμάτευσης προς όφελος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Παίρναμε σε άλλα μέλη που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Πρώτη είναι η κυρία Γκροστέτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Μαρινέσκου που δυστυχώς δεν είναι εδώ για την προσπάθεια που έχει καταβάλει για αυτή τη γνωμοδότηση. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι επιθυμούμε ένα προπολογισμό που θα ευνοεί τη βιομηχανική πολιτική και κυρίω την κοινοτομία στο ύψο των φιλοδοξιών μα. Έχω δύο παρατηρήσει. Πρώτον, για την διαστημική πολιτική πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύξουμε τα εμβληματικά μας προγράμματα, το Γαλιλαίο, το Κοπέρνικο, το Εγνός και την κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία επίσης. Αυτό μας ζητείτε στην έκθεση που εμείς ε, ψηφίσαμε για την Ευρωπαϊκή Διαστημική Στρατηγική. Δεύτερον, δεύτερη παρατήρηση αφορά την τελευταία πρόταση της τελευταίας παραγράφου. Εκεί λέει ο κύριος Μαρινέσκου ότι τα προγράμματα στο διαστημικό τομέα δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται από άλλα προγράμματα. Συμφωνώ επί της αρχής, αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε ότι για την άμυνα αυτό μπορεί να ληφθεί υπόψη μετά το 2020, διότι στην πρώτη φάση του προγράμματος άμυνας ε, ξεκινάμε το 2019, 2019-2020. Οπότε αυτό το βιομηχανικό ε, αμυντικό ε, πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί υπό τις συνθήκες που ξέρουμε, δηλαδή γρήγορα. Ήταν ιστορική η συγκυρία που μας επέτρεψε να το υλοποιήσουμε, οπότε δεν είχε προβλεφθεί αρχικά χρηματοδότηση, Οπότε εν μέρη θα χρηματοδοτηθεί από ανακύκλωση χρημάτων, από ε, χρήματα άλλων προγραμμάτων. Ε, εγώ συγγήτρια για αυτό το βιομηχανικό ε, αμυντικό πρόγραμμα ξέρω ότι τα προγράμματα από τα οποία θα αντλήσουμε χρηματοδότηση δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από αυτή την αντλήση. Κατά τα άλλα συμφωνώ απόλυτα για τον κανόνα, για το μέλλον. Παρ' όλα αυτά ήθελα να κάνω αυτή τη διευκρίνηση διότι είναι πολύ σημαντικό αυτό στην έκθεση που θα παρουσιάσω εγώ σε λίγο καιρό από τώρα. Και συμφωνώ τώρα με τους συναδελφούς που λένε ότι ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να συμμετέχουν ε, ενεργά και ότι όλο, ε, πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη και ότι αυτό είναι σημαντικό και μετά το 2020. Ευχαριστώ. Ο Λεβαντόφσκι, παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Πολύ σύντομα. Τρία σημεία. Πρώτον, για τα σχόλια της Επιτροπής Ήτρε. Είναι πραγματικά πολύ αναγκαία αυτά τα σχόλια. Δεύτερον, για τους ίδιους πόρους. Ως συνεισηγητής μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα επιμείνουμε σε αυτό το θέμα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μας αποθαρρύνουν οι αποτυχημένες προσπάθειες ε, των, του παρελθόντος. Εμείς ε, αυτή τη στιγμή με το Brexit ενδεχομένως έχουμε μπροστά μας μια πολύ καλή ευκαιρία Και τρίτον, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε κάθε λόγο να επιδιώκουμε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει για το ΠΔΕΛΤΑΠΗ μετά το 2020 έω τον Μάρτιο του 2019 πριν τις επόμενε ευρωεκλογέ. Ακόμη λοιπόν και αν η Κομισιόν ε, υποβάλλει την πρόστασή της καθυστερημένα τον Ιούνιο του 2018. Είναι πολύ φιλόδοξος αυτός ο στόχος. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι προηγούμενες ε, διαπραγματεύσεις μας πήραν 2,5 χρόνια και τώρα θέλουμε την ίδια δουλειά να την ολοκληρώσουμε μέσα σε 7 μήνες. Μιλάμε για Φόρμουλα 1 δηλαδή. Πρέπει να σας πω, λοιπόν, ότι παρά τις επιφυλάξεις μου, αξίζει να προσπαθήσουμε. Έχουμε μια ατζέντα ηγετών, η οποία προβλέπει ένα τελείως διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Τον Ιούνιο μετά τις ευρωεκλογές προβλέπεται να γίνει συνάντηση ε, συνδιαλλαγής, ούτε καν δηλαδή οριστικής διαπραγμάτευσης. Έχουμε, δύο διαφορετικά, έχουμε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα, δηλαδή αναθεσμικό όργανο, συμβούλιο και κοινοβούλιο. Ενώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να, υπάρχει ένα κοινό χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστούμε κύριε Λεβαντός και κύριε Σκέλη. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με αυτό που είπαν οι συνάδελφοι νωρίτερα. Είναι πολύ θετικό και η προσέγγιση που περιγράφηκε. Ο κ. Μαρινέσκο έχει κάνει προφανώς πολύ καλή δουλειά και συμφωνώ σε γενικές γραμμές με τις προτεραιότητες που ε, εμφανίζονται εκεί. Σε σχέση με το ζήτημα των ιδίων πόρων και αυτά που είπε ο κύριος Λεβαντόφσκι, γιατί απορρίφθηκε ε, στο παρελθόν. Εμείς δεν συμφωνούμε ούτε αποδεχόμαστε αυτή την απόρριψη, διότι κάθε χρόνο ε, καθίστεται όλο και πιο πρόφυλο το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ίδιους πόρους. Αναφερθήκαμε στο roaming, στο φθηνό ίντερνετ, στα διαστημικά προγράμματα, Κοπέρνικος, Γαλιλαίο κτλ. κτλ. Θα μπορούσε κανείς να αναφερθεί και στο Εράσμους και στο Ταμείο Λιλεγγύης. Όσα περισσότερα λοιπόν μπορούμε να διαθέσουμε σε αυτά τα πολύ αποτελεσματικά προγράμματα, τόσο πιο αποδοτικά θα είναι, τόσο περισσότερο οι πολίτες μας θα αντιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως κάτι θετικό. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο αποφεύγουν όλοι να αναφέρουν. Brexit, πώς θα επηρεάσει τον προπολογισμό, δεν το ξέρουμε ακόμη θα έχει ολοκληρωθεί το Brexit έως ότου ξεκινήσει η νέα ε, δημοσιονομική περίοδος ή θα υπάρξει κάποια παράταση. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι παράγοντες, τις οποίους ε, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, ωστόσο πρέπει να ε, δουλέψουμε με τους παράγοντες που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας και να πείσουμε και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το δικό μας έργο αποβαίνει προς δικό τους όφελος για εκείνους εργαζόμαστε. Και πάλι λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια καλή και γρήγορη αρχή πάντοτε στη βάση των αρχών ώστε να επιτέχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Και νομίζω ότι έτσι θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε κύριε Κέλ. Ξαναδίνω το λόγο στον κύριο Ήλαν για, να... για τις καταληκτικές του παρατηρήσεις παρότι είναι δύσκολο να σας πω ακριβώς αυτά που θα έλεγε ο κύριος Μαρινέσκου. Αυτό στο οποίο συμφωνούμε όλοι πιστεύω. Δεν άκουσα τίποτα ουσιαστικά που να μην είναι κοινή θέση και που να μην μπορούμε να λάβουμε υπόψη. Τα όσα ακούσαμε εδώ ε, βασίζονται σε πράγματα που έχουμε αποφασίσει σε άλλες εκθέσεις. Ουσιαστικά μπορούμε να δεχθούμε όλα όσα ακούσαμε. Απλά να προσθέσω δύο σημαντικά πράγματα και επίσης ξέρω ότι ο κ. Λεβαντόφσκι έχει μια πολύ ρεαλιστική άποψη ε, από τις διαπραγματεύσεις. Δεν πρέπει, δεν πρέπει να ξεκινάμε λέγοντας ότι μπορεί να είναι σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης κάτι και γι' αυτό το λόγο πρέπει να κάνουμε αυτό. Πρέπει να δηλώνουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν αποφασίσει να δαπανούν το 3% του ΑΕΠ και ότι αποτύχαμε και ότι πολιτικά εκεί βασιζόμαστε. Δεν θέλουμε δηλαδή περισσότερο προϋπολογισμό, αν είχαμε πει 20 εκατομμύρια θα... ήταν εντάξει, αυτό θα είχαμε συμφωνήσει. Όταν λέμε 3% δαπάνη του συνολικού ΑΕΠ για έρευνα και ανάπτυξη, εννοούμε ότι δεν αρχίζουμε να μιλάμε σαν να είμαστε ζητιάνοι, μιλάμε βάσει πραγμάτων που έχουμε συμφωνήσει ήδη και λέμε ότι αν δεν γίνει αυτό θα αποτύχουμε. Θα αποτύχουμε. Το δεύτερο, για όσα επικριστούμε. Για να έχουμε τη μετάβαση από έρευνα και καινοτομία σε μεγάλα ε, έργα, θα ζητήσω από τους συντονιστές ε, να σκεφτούν ε, λίγο και την απόφαση που έλαβαν να μην συγκερούν όλη την πολιτική ε, αυτή της ε, Κομισιόν για τη Βιομηχανία ε, θα ήταν λάθος κινήσει. Εδώ είμαστε Επιτροπή Βιομηχανίας. Αν η Επιτροπή Βιομηχανίας δεν πρέπει να συμφωνήσει γνώμη με το έγγραφο το σχετικό της Κομισιόν και να αντικατοπτρίζουν τα όσα λέμε τα διάφορα έγγραφα για τη βιομηχανική πολιτική. Οπότε κάνω μια παράκληση να ξανασκεφτούμε πώς θα ενισχύσουμε κάπως την ε, θέση της Ήτρε χωρίς να παραβλέπουμε, μη παραβλέποντας λοιπόν τα όσα έχει ε, ε, αναφέρει η Κομισιόν να γράψει, δηλαδή ο Πρόεδρος στην Κομισιόν ε, και να της λέει ότι το έγγραφο που έχει δημοσιεύσει είναι το πιο ανεπαρκές που έχουμε δει. Τελικά, όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, πρέπει να λαμβάνουμε τα πάντα υπόψη συστηματικά. Είμαστε επιφορτισμένοι με το EIT, το οποίο δεν αναφέρθηκε. Πρέπει λοιπόν συστηματικά να το εξετάζουμε όλο αυτό, όχι απλά να διαλέγουμε διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι δίνουμε έμφαση σε συγκεκριμένα πράγματα. Βάσει όσο να άκουσα από του συναδέλφου, ε, θέλουμε να καλύψουμε όλε τι πτυχέ, ε, τι δημοσιονομικέ πτυχέ ε, που αφορούν την Επιτροπή Ήτρε και το θεματολογιό της. Οπότε, εν ονόματι του εισηγητή, ζητάω όχι απλά να εστιαστούμε σε ένα ή δύο θέματα, να καλύψουμε όλα τα θέματα για να μην δώσουμε την εντύπωση ότι επιλέγουμε κάποια πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Έλε. 14 Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το σημείο της τη διάταξη. Τελευταίο σημείο τώρα, τα διάφορα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι. Ιδάλλως να κλείσουμε 27 και 28 Νοεμβρίου η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.